Ενημερώνω τους συναδέλφους ότι μετά από την ψηφοφορία θα υπάρχει δυνατότητα έτσι να βγάλουμε μια οικογενειακή εντό εισαγωγικών φωτογραφία εδώ μπροστά από το Προεδρείο. Οπότε σας προσκαλώ όλους εδώ να μείνετε εδώ για να βγάλουμε τη φωτογραφία και στις 6 η ώρα θα έχουμε έτσι μια μικρή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ε, ελπίζω να λάβατε όλη την πρόσκληση. Ε, έτσι, για να ευχαριστήσουμε όλοι ο ένας τον άλλον, αλλά ειδικότερα και τη γραμματεία μας για την εξαιρετική δουλειά που κάναμε. Στο uh, Member Salon G, έτσι, στο ισόγειο θα συναντηθούμε στις 6. Μια μικρή δεξίωση εκεί κοπτά. Αλλά τώρα, αν δούμε... Επιτρέψτε μου απλώς να τελειώσω, συνάδελφο, και θα σας δώσω το λόγο. Εάν λοιπόν δούμε ε, το, τον αριθμό των ψηφοφοριών που έχουν προβλεφθεί για σήμερα αλλά και για την επόμενη Ολομέλεια θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με το αποτέλεσμα ιδιαίτερα μακρόχρονων εδώ τριμερών διαλόγων οπότε πραγματικά ήταν πολύ αποτελεσματικά ε, και πολύ θετικά τα όσα επιτύχουμε και νομίζω πως κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τόσους ε, πολλούς νομοθετικούς φακέλους, τόσα ζητήματα σε τόσο σύντομο διάστημα. Οπότε σας ευχαριστώ όλους και τη γραμματεία που καταφέραμε να το επιτύχουμε. Δίνω τώρα το λόγο στον Φίλιπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ και την οικογενειακή φωτογραφία αλλά επειδή ο δικός μας ε, συντονιστής απουσιάζει, εμείς δεν μπορούμε ως ε, απλοί, αν θέλετε, ευρωβουλευτέ, χωρί το συντονιστή μα να συμμετάσχουμε στη φωτογραφία. Οπότε σα ζητώ συγγνώμη, αλλά εμεί δεν θα ε, είμαστε παρόντε. Καλώ. Ε, δέχομαι λοιπόν τους, ε, το καταστατικό και του ιστορικούς κανόνε τη πολιτική σα ομάδα. Εγώ νόμιζα ότι όλοι οι ευρωβουλευτέ είναι ίσοι, αλλά εντάξει, θα κάνετε αυτό που νομίζετε. Ή μπορούμε με Photoshop να προσθέσουμε το συντονιστή σα μετά στη φωτογραφία. Ο Στάλιν χρησιμοποίησε πιο απλά εργαλεία να το επιτύχει. Λοιπόν, περνάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Έτσι έχουμε λοιπόν αυτήν την ε, τον σχετικό κανονισμό και θα πρέπει να κάνουμε μία ακόμα δοκιμαστική ψηφοφορία γιατί βέβαια τώρα είμαστε μόνο τα μέλη τη Επιτροπή Έγων και χωρί την Μπάτζ. Άρα λοιπόν ξεκινάει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε όλοι. Έχετε ψηφίσει όλοι. Πάντα δοκιμαστική η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Ωραία. Πρώτη λοιπόν ψηφοφορία. Πανεξέταση στο ΕΖΑ. Εδώ ήταν ε, θαύμα σχεδόν το ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα εγκαίρως και όλα τα τμήματα. Οπότε θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Σότ Μαρκάρα και την ε, συνάδελφο Πρέμαν Τσεμπέρες ε, και όλους τους κύριους Οπότε ξεκινάει η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία. The vote 28 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές, εγκρίνεται. Επόμενο. Δύο μάλιστα σημεία που αποτελούν μέρος του ίδιου ε, πακέτου. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται λοιπόν με 28 ψήφους υπέρ, και πέντε κατά λέει ο πρόεδρο, μάλλον εννοεί αποχέ. Περνάμε στο επόμενο τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. This is the ESRB. E λοιπόν το επόμενο. Ah, okay. Vote is closed. Πέρασε η ψηφοφορία και πάλι λοιπόν την ίδια πλειοψηφία των ψήφων υπέρ. Έχουμε συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο που είναι επενδυτικές επιχειρήσεις, investment firms, προληπτική εποπτεία μάλλον των επιχειρήσεων επενδύσεων. προληπτικές απαιτήσεις λοιπόν το πρώτο κομμάτι, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση Πέρασε ψηφοφορία. Ε, εγκρίνεται. Εποπτεία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση is closed. ψηφοφορία, εγκρίνεται και αυτό το κομμάτι. Ε, συγχαίρουμε τον συνάδελφο Μάρκος Φέρμπερ και όλη την ομάδα που συμμετείχε. Περνάμε στα καλυμμένα ομόλογα. Περνάμε στην πρώτη οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα, άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. 29. Η πέραση της ψηφοφορίας, λοιπόν, 29 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Κανονισμός τώρα για τα καλυμμένα ομόλογα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη closed. 29 ψήφοι υπέρ, 4 ε, ψήφοι κατά και 2 αποχές. Συγχαίρουμε τον Μπεντ Λούκε και την ομάδα που διαπραγματεύτηκε. αεφόρες επενδύσεις ε, και γνωστοποιήσεις ε, άρχεται η πάντοτε ονομαστική ψηφοφορία. Vote closed. Πέρας της ψηφοφορίας, 33 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον Πολ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ομοφωνία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα, Ντανούντα, Χίπνερ, CCP. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is ψηφοφορία 29 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 3 αποχές. Συγχαίρουμε την Ντανούτα. Πρόκειται για έναν ακόμα πολύ σημαντικό φάκελο εδώ, να μπαίνοντα υπόψη και το ευρύτερο πλαίσιο. Σβέν Γκίγκολ τώρα, φυσκάλη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία, 30 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και 4 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Την οδηγία για τα NPL για να μην εξυπηρετούμε δάνεια θα την αναβάλουμε για να ψηφίσουμε από τον δύο νόνο ψήξεων καταρχήν. Και έχουμε και την ε, καταρχήν το πρώτο από τα δύο έλληνων non-objection για τις συμβάσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το CCP. Η αλλαγή δηλαδή η οποία απαιτείται λόγω της αλλαγής της ημερομηνία της δυνητικής εξόδου του ΗΠΑ βασιλιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομαδική ψηφοφορία λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην δεύτερη ομαδική ψηφοφορία, τα citations υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συλλογική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τι εκλογέ σκέψης υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Vote is closed πέρασε τη ψηφοφορία 32 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχέ. Δεύτερο τώρα κομμάτι του early non-objection σε ό,τι αφορά ε, την ε, θέση σε ισχύ τη ε, ημερομηνία καθάριση, σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο είδο συμβάσεων. Πρώτη ομαδική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τα άρθρα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Citations. Ομαδική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται ομαδική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τη λογική σκέψη υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται και ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου ονομαστικά ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. The vote is closed. 32 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχέ. Ολοκληρώσαμε και με αυτό το κομμάτι και κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα δύο λεπτών πριν από την τελευταία ψηφοφορία, γιατί πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο εδώ του καταλόγου ψηφοφορίας και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Οπότε για δύο λεπτά διακόπτουμε τις εργασίες μας. Βέβαια.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

Εκ μέρους και του συνεισηγητή συνάδελφοι να σας ενημερώσω σε σχέση με αυτό το τελευταίο σημείο, δηλαδή ε, η οδηγία σε ό,τι αφορά ε, τις ε, επιστοτικές υπηρεσίες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να σας ενημερώσω λοιπόν ως προς το εξή. Μετά από τις ε, εντατικέ διαπραγματεύσει τι οποίε έλαβαν χώρα και προκειμένου να λάβουμε υπόψη μα και τη θέση των υπολείπων πολιτικών ομάδων, κάναμε μία πρόταση η οποία προβλέπει ε, μια αλλαγή ε, όχι μόνο στις ιδεολογικές σκέψεις αλλά και στα άρθρα σε ό,τι αφορά τη λήψη ορισμένων ε, μέτρων η οποία ωστόσο ως αλλαγή δηλαδή μόνο στις ιδεολογικές σκέψεις θεωρώταν ως ανεπαρκής και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη πλειοψηφία έτσι ώστε να περάσουμε στο τριμερή διάλογο. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγικό. Δηλαδή να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτό το κείμενο στο οποίο καταφέραμε να καταλήξουμε σε τόσο θετικό κλίμα και τόσο συναδελφικά αν θέλετε. Οπότε προτείνουμε να μην λάβει χώρα αυτή η ψηφοφορία και να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, εφόσον βέβαια μας το επιτρέψει η πολιτική κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του να μην επιτρέψουν την έγκριση ενός πολύ καλού νομοθετικού κειμένου. Ε, αφήνοντας δηλαδή το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει από αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω πως εδώ τίθεται ένα ερώτημα ως προς τη σοβαρότητα που θέλουν να επιδείξουν οι διάφορες ε, πολιτικές ομάδες. Εάν δηλαδή κανένας δεν είναι διατεθειμένος να είναι διαλλακτικός, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το να έχουμε ένα κακή ποιότητα σε κείμενο. Ας μην αποφασίσουμε το. Ας αναβαλούμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία και ας γίνουν οι διάφορες σωστικές στις πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να δούμε αν μπορεί να λάβει χώρα ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Έστερ βλέπω πως ζητάς το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλά να γραφτεί στα πρακτικά ότι πραγματικά προσπαθήσαμε, παρότι είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και παρά το γεγονός ότι και οι δύο συνεισηγητές θέλησαν να υιοθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις από τις πολιτικές ομάδες, να καταγραφεί παρακαλώ στα πρακτικά ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες προσπαθούμε να βρούμε διατύπωση που είναι σημαντική για μία κυρίως πολιτική ομάδα, αλλά και για κάποιες άλλες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εκείνες τις ε, πολιτικές ομάδες ε, για τις οποίες ε, η διατύπωση στην οποία καταλήξαμε είναι σημαντική. Τις ευχαριστώ λοιπόν για το πνεύμα συνεργασίας, επίσης για την προτιμία που επιδεικνύουν ότι αν γίνουν παραχωρήσεις θα υπερψηφίσουν και θέλω επίσης να καταγραφεί ότι παρότι μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα έκανε τρεις-τέσσερις παραχωρήσεις παρόλα αυτά να ακούει αυτή η πολιτική ομάδα ότι θα καταψηφίσουμε οι υπόλοιποι. Ε, καταλαβαίνετε, αυτό εμένα μου δημιουργεί ερωτήματα κατά πόσον και αυτές οι παραχωρήσεις θα παραμείνουν εάν τελικά ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε με βάση το κείμενο που έχει κατατεθεί, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά, να ευχαριστήσω την Άλντε, ε, την πολιτική ομάδα ESR, το EFDD, την πολιτική ομάδα, η οποία στην ε, τελευταία τελευταία συνεδρίαση δεν ήταν 100% ε, φτυχισμένη, αλλά τουλάχιστον επέδειξαν πνεύμα συνεργασία. Ευχαριστώ και την Κούε για την ε, ανοιχτή συνεργασία που βοήθησαν και άφησα μία συγκεκριμένη ομάδα ξέρετε όλοι ποια είναι, η οποία θέλει όλο και περισσότερες παραχωρήσεις ε, σε, αυτές τις διαπραγματεύσεις και τελικά τι κάνει, καταψηφίζει και αυτή υποτίθεται ότι αυτή είναι και το κέντρο της πολιτικής ε, στην Ευρώπη. Υποτίθεται είναι στο κέντρο και θέλει ε, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να αντιμετωπίσει όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες. Ε, εγώ δεν τα βρίσκω σωστά αυτά. Για όλους τους άλλους ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Έστερ. Μισό λεπτό, θα σας δώσω το λόγο. Ε, πράγματι, θα καταγραφεί στα πρακτικά και είναι απόλυτα σαφές ότι αν τελικά συγκρίνουμε το πώς έχει η κατάσταση. Αν δούμε πώς έχει η κατάσταση, ε, με το κείμενο θα αυξηθεί κατά πολύ η προστασία του καταναλωτή. Αν δεν υπάρχει κείμενο, επειδή ε, δεν συμφωνούν κάποιες πολιτικές ομάδες, πάμε πάλι πίσω εκεί που είχαμε ξεκινήσει, άρα δηλαδή ε, αυτό πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά για να ξέρουμε ποιος φταίει και γιατί δεν μπόρεσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο Βέρνερ έχει τον λόγο. Κοιτάξτε, αυτό αποτελεί απόδειξη για το γεγονό ότι κατά την επόμενη θητεία πρέπει να επανεξεταστούν οι κανόνε. Όταν λοιπόν έχει ψηφίσει η Ολομέλεια ε, και το μόνο που απομένει είναι η τελική ψηφοφορία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει. Αν όμω με βάση την ψηφοφορία στην Επιτροπή και τη συμπεριφορά ε, οκτώ ατόμων γίνονται τέτοια βήματα, τότε το μόνο που μπορεί να γίνει είναι και με τέτοιου είδου δύσκολα θέματα να πηγαίνει πηγαίνει κανείς στην αλλομέλεια. Μετά πια δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα. Για μένα αυτό είναι ένα μάθημα που εξάγω από τη συμπεριφορά των πρασίνων. Ο κύριος ε, Λούκε έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να γραφτεί στα πρακτικά ότι εγώ ε, και το σύνολο της πολιτικής ομάδας, το ECR, ε, τα υπερψηφίζαμε σήμερα γιατί είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα αυτό το οποίο ε, κατατίθεται, αλλά το να αποδίδουμε όλη την υπετιότητα στους πράσινους νομίζω ότι δεν είναι και σωστό γιατί ξέρετε υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση και οι σκιώδεις ε, είχαν τεράστια πίεση. Είχαμε μόνο μία συνάντηση σκιωδών, δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε όλες τις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις και ένα τέταρτο νωρίτερα από το τέλος ε, προτάθηκαν νέες διατυπώσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα τελικά να έχουμε λίγο χρόνο τα εξετάσουμε αυτά και να δούμε ε, κατά πόσον αυτά που θα αποφασίσουμε το όντι κατά πόσον έχουν βάση. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρος. Πράγματι, είναι πρόβλημα αυτό αν υπάρχει πίεση χρόνου και γι' αυτό να βάλουμε. Άρα δηλαδή την επόμενη εβδομάδα πράγματι όλες οι πολιτικές ομάδες θα έχουν το χρόνο να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο. Ο Φίλιπ. Ε, ορισμένοι από εσά μιλάτε για την ομάδα της οποίας, την οποία προεδρεύω. Αισθάνομαι υποχρεωμένο να πω δύο λόγια. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε ε, του φακέλου, δεν μπορώ να μιλήσω επί τη ουσία. Συμφωνώ με αυτού που είπαν ότι συνήθω, όταν γίνονται παραχωρήσει ως τμήμα μέσα στα πλαίσια της συνολικής, του συνολικού παζαρέματο, ο καθένα θα πρέπει να τηρήσει τι δικέ του δεσμεύσει. Δεν ξέρω τι φύση είχαν οι συζητήσει από αυτά που ξέρω είναι ότι εγώ πάντα ξεκαθαρίζω από την αρχή εάν συμφωνώ με, την, με το παζάρεμα αυτό ε, και τη συμφωνία και την τηρώ. Αλλιώς δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω τι υπόθηκε από τους εισηγητές. Άκουσα τι είπατε. Αλλά ο εισηγητής δεν είναι εδώ και δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Φαντάζομαι ότι η συνολική ισορροπία δεν είναι ικανοποιητική και συμφωνώ ότι όταν κάνει κανείς ε, παραχωρήσεις για να συμφωνήσουν όλοι ε, και παρόλα αυτά δεν συμφωνούν, τότε αυτές οι παραχωρήσεις δεν ισχύουν πια. Λογικό. Το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως ε, είναι ότι η συνολική ισορροπία δεν είναι ικανοποιητική, αλλά δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν ξέρω το θέμα αρκετά. Κατέγραψα πάντως αυτά που είπατε. Σου. Πολύ ωραία. Ο κύριος Τρεμόζα. 30 δευτερόλεπτα. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο κάναμε μια πολύ χρήσιμη συνάντηση σκιωδών. Εγώ παρουσίασα 31 τροπολογίες και 25 συμπεριλήφθηκαν συμφωνία. Και το ίδιο νομίζω να συμβαίνει και για τους πράσινους. Οι δύο συνεισηγητέ κάνουν μια πολύ καλή δουλειά στη δική μου περίπτωση και είναι κρίμα που ο σκιώδη συζητητή σα δεν είναι εδώ, γιατί στις εκλογές θα ακούσουμε και θα διδαχθούμε, θα λάβουμε πολλά ηθικά διδάγματα για αυτές τις νέες πολιτικές. Είναι πολύ σημαντική χρονική στιγμή και είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι σκιώδη εισηγητές. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να τα πω αυτά δημόσια. Ε, εμείς δεν δίνουμε μαθήματα στους άλλους, εμείς οι πράσινοι, έτσι. Εντάξει. Όσοι δεν ξέρουν το κείμενο δεν μπορούν να ερμηνεύσουν πολύ καλά τα τη συζήτηση. Το καταλαβαίνω. Θα συνεχίσουμε πάντως τις συζητήσεις. Την επόμενη Πέμπτη έχουμε τελευταία ευκαιρία να ψηφίσουμε για αυτό το θέμα. Τα... Οι βουλευτές μπορούν να πάνε στην δεύτερη σειρά 16 με 22 για την ε, φωτογραφία μας. Κλείνει εδώ η συνεδρίαση.